Ξεκινάει λοιπόν η συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας κάνω μία ανακοίνωση. Εκτελώντας ε, μία απόφαση της, ε, του Ιταλικού κράτους, ε, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο στη συνεδρίασή του στις 6 Ιουνίου 2011 ανακήρυξε ως εκλεγέντα με τον κατάλογο του κόμματος Popolo della Libertà στην Βόρεια Ιταλία τον κύριο Τζουζέπε Γκαργάνη, που εγκατιστά τον κύριο Τζοβάνι Γκολίνο, του οποίου η θέση εντάσσεται στον κατάλογο της ε, Ανατολικής Ιταλίας. Και ε, αυτό ισχύει, η πράξη αυτή ισχύει από τις 6 Ιουνίου 2011. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον συνάδελφο. Τα πρακτικά της ε, χτεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν διανεμήθηκαν. Εάν έχετε παρατηρήσεις παρακαλώ να τις ε, εκφράσετε τώρα. Αν όχι, ε, τα πρακτικά ε, θεωρώ ότι έχουν πλέον εγκριθεί. Η μερίσια διάταξη προβλέπει τώρα τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το Ουγγρικό, αναθεωρημένο Ουγγρικό Σύνταγμα. Και θα ήθελα ευθύ αμέσω να δώσω το λόγο στον, στην κυρία Γκιόρη στην Υπουργό κυρία Γκιώρη. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, αξιότιμα μέλη. Η συνθήκη δεν έχει μεταβιβάσει στο Συμβούλιο καμία εξουσία να ασχολείται με τα εθνικά